προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας όσον αφορά την κατάσταση στο Μπουρούντι. Ο Επίτροπος Σταυροβιτς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, όπως ξέρετε, έχουν γίνει πολλέ συζητήσει και έχουν εγκριθεί πολλά ψηφίσματα για τον Μπούροντα του τελευταίου μήνε. Πιστεύω όμω ότι τα τελευταία σοβαρά γεγονότα στη χώρα δικαιολογούν πλήρω το να συζητήσουμε αυτό το θέμα ξανά σήμερα το απόγευμα. Όπω είπε και ο Επίτροπο Μίμητσα όταν απευθύνθηκε στο Σώμα τον Απρίλιο, είναι σημαντικό ε, οι κάτοικοι του Μπουρούντι να ξέρουν ότι η φωνή του ακούγεται και στην Ευρώπη για να έχουν ε, ε, την πιθανότητα η δημοκρατία της χώρας τους να είναι ανθεκτική και να γνωρίσει μακροζωία. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών της χώρας αυτής, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους. Έχουν ε, υπάρξει πολλέ εξελίξει μετά από τι τελευταίε συζητήσει στο σώμα αυτό στη χώρα του Μπουρούντι και αυτό ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξέρετε ότι η απόφαση του κυβερνητικού κόμματο να ορίσει τον ε, πρόεδρο Γκουρούνζιζα ω ε, ως, ε, υποψήφιο του το προεδρικό αξίωμα δημιούργησε διχασμό στην κοινωνία τη χώρα. Η κατάσταση ε, επιδεινώθηκε ε, πολύ γρήγορα με την απόπειρα πραξικοπήματος στις 13 Μαΐου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πραγματικά καταδικάζει κάθε πράξη πολιτικής βίας. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να ενθαρρύνουμε την ε, ανοιχτή τη ε, προσέγγιση και την διαφάνεια που πρέπει να ακολουθεί στον Μπουρούντι για να υπάρξει συμφιλίωση και σταθερότητα στη χώρα. Προφανώ η διεθνή κοινότητα, ε, συμπεριλαμβανομένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει μια κατάσταση πολύ ε, ανησυχητική. Όπω η αντιπρόεδρο, είπατε εκπρόσωπο Μογκερίνη, είπε στη δήλωσή τη μετά τα γεγονότα τη 14η Μαου, οι πρώτε μα σκέψει πρέπει να, προς τους, να κατευθυνθούν προ του πολίτε τη χώρα, την ασφάλεια και την ε, του ε, προτού η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι ανησυχίε αυτέ αφορούν και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Από την ανθρωπιστική άποψη και εφόσον η πολιτική κρίση ξέσπασε στο Μπουρούντι, στο Μπουρούντι είναι, είναι χιλιάδε οι πολίτε που ε, φεύγουν από τη χώρα μαζικά τι τελευταίε εβδομάδε. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν ξεφύγει στι γειτονικέ χώρε, την Τανζανία, τη Ρουάντα, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Υπηρεσία για την Προστασία των Πολιτών παρακολουθεί στενά την κατάσταση και Ήδη έχει προβλεφθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις άμεσες ανάγκες των προσφύγων από τον Μπουρούντι που φτάσαν την Ρουάντα μόλις τον τελευταίο μήνα. Επιπλέον, ανθρωπιστική βοήθεια προσφέρεται ε, για τις ειδικέ ανάγκες των προσφύγων που έχουν φτάσει στην Τανζανία ε, καθώς ε, και για την αντιμετώπιση επιδημιών, ασθενειών και ενδεχομένως για χολέρα. Ε, την περίπτωση κρούσματων χολέρας. Χρειάζεται όμως και πολιτική δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον Μπουρούντι στις προσπάθειες να θεμελιώσει τη δημοκρατία της μετά ε, τα, την πάυση των χροπαξιών και του εμφυλίου πολέμου. Η χώρα πρέπει να περάσει σε μια νέα εποχή. Οι νομοθετικές και προειδικές εκλογές ήταν ένα καθοριστικό βήμα για να ε, η δημοκρατική όψη της ε, του καθεστώτο του Μπουρούντι. Γι' αυτόν τον λόγο, είπατε, εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο Μογκερίνη αποφάσισε να αποστείλει ε, αποστολή ε, παρατήρησης των προεδρικών εκλογών με επικεφαλή τον Ευρωβουλευτή David Μάρτιν. Εδώ πρέπει να ε, επενέσω τον κύριο Μάρτιν για την αφοσίωσή του και την, τον ζήλο του κατά τις δύσκολες αυτές αρμοδιότητες που ανέλαβε. Ε, Επίση, η ειρηνευτική συμφωνία και η τήρησή τη είναι καθοριστική σημασία για τη σταθερότητα στη χώρα. Αυτή είναι η πρωταρχική αρχή την οποία όλοι θα πρέπει να σεβαστούμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό βρίσκεται στην ε, καρδιά της σύραξης και ότι ε, θα πρέπει και ο πρόεδρος της χώρας να κληθεί να σεβαστεί πάνω από όλα τα συμφέροντα της χώρας. Για να πετύχουν οι εκλογές θα πρέπει να υπάρξει ευρεία συνένεση για τα θέματα αυτά. Το να υπάρξει λοιπόν αποστολή για την παρατηρήση των εκλογών και ε, να στηρίξουμε την ε, νόμιμη διεξαγωγή τους έχει να κάνει με την ειρηνική αξιόπιστη και δίκαιη μεταχείριση όλων των πολιτικών φορέων και συμμετεχόντων στις εκλογές ως ψήφοι. Ε, θα πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα στις εκλογές. Αυτό είναι ο στόχος μας, αλλά για να το πετύχουμε πρέπει να ε, πληρώνονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Δυστυχώς η αποτίμησή μας είναι ότι οι προϋποθέσεις αυτές για την ώρα δεν μπορούν να πληρούνται. Ε, κυρίως γιατί βλέπουμε διαρκώς να πολλαπλασιάζονται οι περιορισμοί στα ανεξαρτά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην ελευθερία έκφρασης και την άσκηση βίας κατά των διαδηλωτών, αλλά και το κλίμα εκφοβισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, με την έλλειψη της εμπιστοσύνης στις ε, αρμόδιες αρχές να εντείνεται. Οι εξελίξει των τελευταίων ημερών και το περασμένου μήνα ε, ενισχύουν αυτές τις ε, ανησυχίες μας. Για αυτό το λόγο αναστήλαμε την αποστολή για την παρατήρηση των εκλογών και δεν θα μπορέσουμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας προς τις εκλογές αυτές. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε για την αξιοπιστία των εκλογών την περασμένη εβδομάδα Ελλάδα Δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παρετήθηκαν η Αφρικανική Ένωση και η κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής απόσχουν από το να, αποστήσουν, να αποστείλουν ε, αποστολή για την παρατήρηση των εκλογών στον Μπουρούντι. Αλλά δεν τελειώνει εδώ το όλο πρόβλημα. Οι εθνικοί εταίροι στον Μπουρούντι θα πρέπει να συμφωνήσουν να οργανωθούν ε, δημοκρατικές εκλογές. Τότε ευχαρίστως να αποστείλουμε την αποστολή όπως έχει οργανωθεί και να τους υποστηρίξουμε και θα πρέπει οι προποθέσει αυτέ να εκπληρώνονται. Οι όροι αυτοί να πληρούνται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν γύρω από ένα τραπέζι διαλόγου για να βεβαιωθούν ότι ε, τηρούν του ίδιου κανόνε και θα πρέπει η κυβέρνηση του Μπουρούντι να επιτρέψει σε όλου του ε, φορεί τη χώρα να εκφραστούν ελεύθερα με επόμενη τι αρχέ τη δημοκρατία. Η ε, Δημοκρατική Ένωση θέλει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στην πολιτική κρίση στο Μπουρούντι. Ε, υπό το φως ε, των αποφάσεων της κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής, της Αφρικανικής Ένωσης και της ε, ευρύτερης περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Αφρικής. Όπως ξέρετε η Αφρικανική κοινότητα συνέκαλε, συνεκάλεσε στον Ντάρεν Σαλάμ μια έκτακτη σύνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Και να μην ξεχνάμε τα πορίσματα της σύνοδο αυτή. Διότι στηρίζουν, θα καθορίσουν τα πορίσματα αυτά την δική μας πορεία για τις ερχόμενες εβδομάδες. Πρέπει η Αφρικανική ε, κοινότητα, να πούμε ότι η Αφρικανική κοινότητα ε, αναγνώρισε το έργο του κυρίου Τζένιντ που είναι ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ για τα θέματα της ε, Ανατολικής Αφρικής. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μας και ελπίζουμε ότι οι προσπάθειές του θα ευοδοθούν ώστε όπως είπε και ο εκπρόσωπος της κυρίας Μογκερίνη στις 3 Ιουνίου, ε, θα έρθουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, γύρω από ένα τραπέζι διαλόγου με συμμετοχή της κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής και των εκπροσώπων της Αφρικανικής Ένωσης για να βρούμε μια συνένεση για την πορεία που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση περιφερειακά και μετά και διεθνώς κατά προτεραιότητα. Στηρίζουμε την προσπάθεια της κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής να αναπληθούν οι εκλογές και σημειώνουμε ότι σήμερα μόλις ένα προεδρικό διάταγμα ορίστηκε ορίζοντας ένα νέο πρόγραμμα πρόγραμμα για τι εκλογέ, ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Όμω αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν θα μπορέσει να τηρηθεί εφόσον δεν συνοδευτεί από ταχύ και σοβαρέ προσπάθειε να επιτευχθεί η, συνένωση, η συνένεση και να υπάρξουν τα απαραίτητα βήματα προ την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα συμπεράσματα τη Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να συνοδευτούν από χειροπιαστέ δράσει. Την πάυση τη άσκηση βία από όλε τι πλευρέ και τον αφοπλισμό των ε, ένοπλων ε, νέων και ανταρτών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βεβαιωθεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίε ε, γίνονται σεβαστά. Η κυβέρνηση του Μπουρούντι θα πρέπει αυτέ τι ε, προποθέσει να τι εξασφαλίσει για να πάψει κάθε μορφή βία. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρήσει τι ε, προθέσει τη μακροπρόθεσμα, όμω θέλω να υπογραμμίσω τι ανάγκε τη παρούσα στιγμή. Το να γίνουν επιτυχημένε εκλογέ δεν θα είναι κάτι το απλό. Θα πρέπει όλοι οι πολίτε πολίτες του Μπουρούντι να στηρίξουν τις προσπάθειες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Αφρικανικής Ένωσης και της ε, κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής για να επικρατήσει ένα ε, ομαλό κλίμα. Το γνωρίζουμε αυτό, ε, γιατί οι ε, πολίτες του Μπουρούντι έχουν δεσμευτεί ε, με τις αρχές αυτές μέσω των συμφωνιών του Κοτονού και για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, καθώς και των κοινοβουλευτικών αξιών. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα έχουμε κατά νου, να αφήσουμε και χώρο στους πολίτες του Μπουρούντι, καθώς και στους περιφερειακούς και τοπικούς τους εταίρους, να βρουν λύση στην κρίση. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντα κάτι σημαντικό. Το είπε ο Επίτροπο Μίμητσα τον περασμένο μήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα σενάρια και να δει κατά πόσο θα χρειαστούν τα μέτρα. Ενδεχομένω και για την αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ τον Μπουρούντι. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν διαφορετικά μέτρα στον πληθυσμό τη χώρα, αλλά και τη σταθερότητα τη χώρα και τη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις των βουλευτών. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις παρεμβάσεις εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Θα δώσω λοιπόν πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Ζέλερ εκ μέρους του ΕΛΚ για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πέτρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σωστό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατ' επανάληψη στρέψαμε και στρέφουμε το βλέμμα μας στον Μπορούντι μετά από αυτό τον ε, πολιτή εμφύλιο πόλεμο με χιλιάδες νεκρούς. Ε, και μετά τις ε, εκλογές, με τις εκλογές ε, η χώρα αυτή η οποία είναι μια από τις φτωχότερες του κόσμου ήθελε να κάνει ένα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ε, των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διατεθειμένη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, έθεσε απελευθέρωση 6 εκατομμύρια και μια ομάδα ήταν διατεθειμένη να συνοδεύσει, να μεταβεί εκεί και να παρακολουθήσει τις ε, εκλογές. Αλλά ε, μετά την ε, προσπάθεια του Προέδρου να υποβάλει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθούν κανονικά οι εκλογές. Ε, υπάρχουν ε, εκατοντάδες ε, χιλιάδες πολίτες του Μπουρούντι που μετά το ξέσπασμα της βίας εγκατέλειψαν τη χώρα και το κόμμα του Προέδρου τρομοκρατεί όλους όσους ε, υποτίθεται ότι είναι ενάντια στο καθεστώς. Ο συμβασμός ο οποίος ε, είχε βρεθεί μεταξύ των εθνικών ομάδων Χούτου και Τούτσι ε, κινδυνεύει να διαλυθεί και εθελοντικοί οργανισμοί της Εκκλησίας αποσύρθηκαν. Η κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής ε, πρέπει στη σύσταση αναβολής των εκλογών, αλλά ωστόσο αυτή η συνάντηση κορυφής δεν έλαβε χώρα ε, ε, δεν έλαβε συγγνώμη θέση εν σχέση με την πρόθεση του Γκουρουνζίζα να υποβάλει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία και επίκενται εκλογές στο Κονγκό και του χρόνου στη Ρουάντα και εκεί θα μπορούσε επίσης οι πρόεδροι των χωρών αυτών εντελώς αντισυνταγματικά να υποβάλουν υποψηφιότητα για μια τρίτη προεδρική θητεία. Πολλοί πρόσφυγες από το Μπορούντι επιβαρύνουν σημαντικά τις κυτερνικέ χώρες, την Τανζανία, τη Ρουάντα και το Κονγκό. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τις ε, χώρες της Αφρικανικής Ένωσης να αναλάβουμε κοινή δράση ούτω ώστε ήδη αυτό το χρόνο να διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές στο Μπουρούντι. Υπάρχουν δυνατότητε άσκησης επιρροής. Θα μπορούσαμε να πάυσουμε την οικονομική βοήθεια προς το Μπουρούντι και να βοηθήσουμε βεβαίως τους ε, πρόσφυγες ε, μέσω διοργάνωσης στρατοπέδων προσφύγων και να υποστηρίξουμε τους πολίτες για μια δημοκρατική διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα αυτή. Κύριε έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Στοβίτς. Στέχεστε. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εσείς τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που σιγά σιγά βγαίνουν από την ύφεση που έτσι καλλιώς πλήγει πολλές γενιές νομίζετε ότι ευχαρίστως θα άκουγαν ότι τα χρήματά τους και ο χρόνος τους πηγαίνουν στο Μπουρούντι όταν αυτοί περνάνε τόσο δύσκολε στιγμέ. Νομίζετε ότι θα χαιρόντουσαν πολύ αν σα άκουγαν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Όπως ξέρετε, ε, ε, πρόκειται για καθήκον των ευρωπαϊκών χωρών να βοηθούν τι αναπτυσσόμενε χώρες και μεταξύ αυτών εντάσσεται, λέγεται και το Μπορούντι εφόσον οι χώρες αυτές ε, προτίθενται να εκδημοκρατιστούν. Αυτό ήταν και ο στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας και γι' αυτό το αίτημά μου ε, μέχρι ότου ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες εκεί να πάυσει η χορήγηση οικονομικής ε, βοήθειας. Ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο ήδη το έχουν πράξει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρτιν τώρα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μίλησαν για 1,5 δισεκατομμύριο προκειμένου να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Καλό αυτό. Η αστάθεια στο Μπουρούντι ε, πράγματι δεν είναι σφάλμα των γειτόνων, δεν θα πρέπει ούτε οι γείτονες να υποφέρουν. Επίσης ευχαριστώ την Επιτροπή για τα σχόλια που έκαναν όσον αφορά τις καλές υπηρεσίες των παρατηρητών. Όταν ήμουν εκεί είδα πόσο πολύ έχει δεσμευτεί και η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να βρούνε λύσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τον Μπουρούντι. Ήμουν εκεί λοιπόν, συζητήσαμε και τις δράσεις βάσει του άρθρου 96. Οπότε πολύ χαίρομαι που έχουμε δεσμευτεί πλήρως στη χώρα. Τώρα όπως είπε και ο Πίτροπος, ο κύριος Ναυράτσης, ο κύριος λόγος της αστάθειας και των ταραχών είναι το ότι ο πρόεδρος προσπάθησε να πετύχει μια τρίτη θητεία. Πρόκειται για παραβίαση των συμφωνιών της Αρούσα και οι συνέπειες της προσπάθειας αυτής ήταν ε, βία στο δρόμο από τους παραστρατιωτικούς, όχι από τους διαδηλωτές, από τους παραστρατιωτικούς που προσπάθησαν να καταστήλουν τις ειρηνικές αυτές διαδηλώσεις στους δρόμους. Και το πρώτο που πρέπει να γίνει στο Μπουρούντι είναι οι επίσημες υπηρεσίες ασφάλειας να παραγωνίσουν τους παραστρατιωτικούς. Αν θέλουμε τώρα βελτίωση στην κατάσταση στο Μπουρούντι θα πρέπει να μπορεί και αντιπολίτευση να κάνει τη δικιά της εκστρατεία. Όταν ήμουν εκεί κατάλαβα ότι οι κυβερνητικές ε, δυνάμεις μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους υποστηρικτές τους, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια της αντιπολίτευσης να έχει κάποιο χώρο να μπορεί να μιλήσει, κάποιο φόρουμ, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να ανοίξουν και πάλι. Και είδα τους πολίτες να βλέπουν ότι δεν μπορούν να έχουν εκπομπές και ότι προσπάθειες ε, γινόντουσαν δεν πετύχαιναν. Από την άλλη η κυβέρνηση λέει είσαστε ελεύθεροι. Συνεπώς οι συνθήκες δεν είναι καλές για να υπάρξουν ε, μέσα ενημέρωσης ελεύθερα θα έπρεπε όμως, και τελειώνω πρόεδρε, στις 29 Ιουνίου με 15 Ιουλίου, αν δεν υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, θα έλεγα να ξαναπάμε στον Μπουρούντι, γιατί προς το παρόν δεν είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρατηρήσει χωρίς πρόβλημα τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μισελ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν πρέπει να συνεχίζουμε να κλείνουμε τα μάτια βέβαια μπροστά στις ταραχές, στο χάος και στις φαγές που γίνονται στον Μπορούντι. Σήμερα καταστράφηκε ανεξάρτητα το ραδιόφωνο, τηλεοπτικά κανάλια που προσπάθησαν να πούν κάτι διαφορετικό. Ορισμένοι έφυγαν από τη χώρα, άλλοι κρύβονται στην παρανομία, διεξορία για μερικούς. Δεν βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση και η αντιπολίτευση Ήδη έχει κυνηγηθεί και είδαμε τις σφαγές 23 Μαΐου. Οι διώξεις λοιπόν οδηγούν σε καταστολή του ίδιου του κράτους δικαίου. Και τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα ότι η εθνικιστική φλόγα ανάβει και πάλι και ξέρουμε σε τι δράμα οδήγησε αυτό την τελευταία φορά. Συμμετείχα το 2001 στις συμφωνίες της Αρούς εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορώ να σας πω ότι η απόφαση να μην συμμετέχει ο πρώτος εκλογές αυτές είναι κάτι εντελώς παράνομο. Για μένα δεν έχει κανένα δικαίωμα να προχωρήσει. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πει ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από εκλογές τέτοιες παράνομες δεν θα αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια τυφλή καταστολή κατά της αντιπολίτευσης. Πρέπει να επιστρέψουν οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης στη χώρα, να ελευθερωθούν χωρίς όρους οι πολιτικοί κρατούμενοι και να πάψει αυτή η όχληση που συνεχίζει κατά της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να τους απειλήσουμε ότι θα κλείσουμε τους λογαριασμούς τους στους τραπεζικούς των υπευθύνων, εκείνων που προβαίνουν σε βία κατά των πολιτών. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο τελευταίος πρόεδρος να συνεχίσει να ζητάει την εντολή του λαού. Δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Αυτό είναι απόλυτο. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βεζιά έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από η τελευταία μας συζήτηση μετά την εξαγγελία του Πρόεδρου Γκουρουνζής να υποβάλει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία η βία αυξάνεται ε, πάρα πολύ. Ε, κάτοικοι είναι νεκροί και άλλοι φεύγουν από τη χώρα ε, ένας ηγέτης ενός μικρού κόμματος της αντιπολίτευσης δολοφονήθηκε και οι άλλοι πολιτικοί βρίσκονται, δρούν παράνομα. Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο χρονοδιάγραμμα το οποίο όμως δεν πρόκειται να ρυθμίσει τα πράγματα και η επιτροπή αυτή έχει χάσει εντελώς το κύρος της γιατί δύο από τα μέλη της έχουν ήδη διαφύγει και θα πρέπει να πάρει αποφάσεις με τέσσερα πέμπτα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, προτάσεις για την διεξαγωγή των ε, νέων εκλογών με τη σύσταση μιας νέας επιτροπής. Οι αρχές του Μπουρούντι ε, υποκρύπτονται πίσω από θεσμικούς λόγους για τους οποίους λένε δεν μπορούν να αναβληθούν πλέον οι εκλογές. Ε, η ε, εκλογική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νόημα ε, θα μπορούσε βεβαίως να μεταβεί εκεί εφόσον εξασφαλιστούν οι συνθήκες διεξαγωγής νόμιμων εκλογών. Αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο εν μέσω αυτής της ε, βίας. Οι αρχές ε, του Μπουρούντι παραμένουν ε, βοβές. Η ισορροπία στην περιοχή απειλείται και υπάρχει απειλή νέας εμφύλιας σύραξης υπάρχει ένα κίνημα βέβαια κατά της κυβέρνησης. Ε, η, χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από, τις, ε, από την ξένη βοήθεια. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 400 ε, εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να στραφούν προς, το, προς τη στήριξη του πληθυσμού και θα πρέπει να αποτρέψουμε μια νέα σφαγή. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στο Μπουρούντι είναι πολύ σοβαρή. Υπόθηκαν ήδη πάρα πολλά πράγματα σχετικά. Ε, είναι το αποτέλεσμα μιας ε, παραμονής στην εξουσία ενός ε, τυραννικού προέδρου. Ε, και ήταν μια επιτυχία η έκκληση της ε, Ανατολικής ε, Αφρικής σε σχέση με την διεξαγωγή των εκλογών. Αλλά η αιμονή του Κουρουντζίζα να υποβάλει υποψηφιότητα θέτει σε κίνδυνο την κανονική διεξαγωγή των εκλογών. Και τώρα απομένει το ερώτημα τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα ε, θα πρέπει να ε, παρατηρήσει τα μέσα, ε, τα θεσμικά όργανα στο Μπουρούντι και θα πρέπει να ε, προσέξει ε, να μην ξεσπάσει το εθνοτικό μίσος όπως ε, στη Ρουάντα μεταξύ των Χούτου και των Τούτσι. Δεν θα πρέπει να ενισχύεται, να το εθνοτικό αυτό μίσος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, υπάρχουν οι παραστρατικές οργανώσεις και οι πολιτοφυλακές ε, οι οποίες ε, προβαίνουν σε πράξεις βίας. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στο Κοτονού. Στο Κοτονού ή για το Κουτονού θα είχαμε τη δυνατότητα, ή μέσω του Κοτονού θα μπορούσαμε να αναστείλουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Το είπε ο κυριο τσελλαρ Ποια είναι η δική σα τοποθέτηση σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα αναστολή τη βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν προβλέπει να προσανατολιστούν τα κονδύλια του προπολογισμού σε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια γιατί χρειάζονται χρήματα για τους μετανάστες και για την καταπολέμηση της χολέρας ή ε, θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για να θέσουμε σε πίεση την ε, κυβέρνηση το, του Μπουρούντι τι πρόκειται να πράξετε πέρα από την παρατήρηση των εκλογών προκειμένου να στηρίξετε τον ε, διάλογο μεταξύ κοινωνίας πολιτών. Και... Ευχαριστούμε ο κύριος Καστάλντο. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε την πολλωστή παρεκτροπή της ε, Αφρικής και το δίλημα του λαού του Μπουρούντι που θυμώνεται ε, στο ραδιόφωνο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, διαδηλώσεις λοιπόν κατά του ε, δικτατορικού Προέδρου, ο οποίος παραβιάζει τις συνταγματικές ελευθερίες, ζητώντας να έχει τρίτη προεδρική θητεία. Ουσιαστικά πρόκειται για πραξικόπημα κατά του κράτους δικαίου, κατά του νόμου, κατά του, των συμφερόντων του λαού του. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία και ο στρατός θα έπρεπε να προστατεύουν ε, την ε, ισορροπία μεταξύ Χούτου και Τούτσι και να μην προκύψει εθνοτική ε, σύραξη που να μοιάζει με την γενοκτονία. Όμως ο, ο πληθωρισμός της χώρας που ξεφεύγει από τον έλεγχο, φυγή των ε, προσφύγων και η δράση του στρατού δεν επιτρέπουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, στην πραγματικότητα, κανένα αξιόπιστο διάλογο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ του κυβερνώντο κόμματο και τη αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη και διχασμένη. Και οι ηγέτε τη Ανατολική Αφρική είναι πολύ αμφίσιμοι και καθόλου ε, συγκεκριμένοι. Πρέπει λοιπόν μόνο να, να δούμε ότι μόνο οι εκτεβιστέ προστατεύουν την κοινωνία των πολιτών και του πολίτε τη χώρα αυτή. Είναι δική μα ευθύνη και δικοί τους να ε, σεβαστούμε, να κάνουμε τα θεμελή δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Θα πρέπει να, ζητηθούν, να ζητηθεί εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος βεβαίως για να θεμελιωθεί το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα αυτή, αλλά πολλές φορές αυτό σημαίνει και απώλεια χρόνου. Και θα πρέπει χωρίς ε, εξαιρέσεις να ζητήσουμε την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων. Εάν ζητηθούν εθελοντές για την ε, αποστολή παρατήρηση των εκλογών, εγώ θα προσφερθώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, πολύ. Do Μπλε κάρτα στον κύριο Μάρτιν. Συμφωνώ με πολλά από όσα Όταν ήμουν όμως στον Μπουρούντι, η, πρώτη, η, μόνη κυβέρνηση προσπαθούσε να μετατρέψει αυτή τη σύραξη σε εθνοτική σύραξη. Πρόκειται για πολιτική σύγκρουση και δεν θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι του. Συμφωνείτε σε αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, ε, και μάλιστα αυτό που είπα προηγουμένω, ήταν ακριβώ αυτό. Δηλαδή οι συμφωνίε τη Αρούσα λειτουργήσαν και η κυβέρνηση προσπαθεί να ε, αναδιαμορφώσει την εθνοτική σύγκρουση για να κρύψει τις δικές της αδυναμίες. Άρα δηλαδή πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε αυτό το παιχνίδι του Προέδρου να βρει την συνένεση και κυρίως ε, για άλλη μια φορά να του επισημάνουμε τις ευθύνες του. Σας ευχαριστώ. Yes, you have a point of order. Yes. Διαδικαστικό θέμα, πράγματι, για το άρθρο, με βάση το άρθρο 191 νωρίτερα. Οι διάφοροι συναλφοί ζήτησαν την διακοπή της ε, Συνόδου ως ε, διαμαρτυρία για τον δυσάρεστο τρόπο με τον οποίο ε, γίνονται συζητήσεις. Πιστεύουμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Τώρα θα θέλαμε να προτείνουμε ένα συμβιβασμό εκ μέρους της ομάδας EFTD. Θα θέλαμε να προτείνουμε να διακοπεί η Σύνοδος για το υπόλοιπο της ημέρας για να μας δώσετε λίγο το χρόνο να σκεφτούμε για τον μη δημοκρατικό, αντιδημοκρατικό τρόπο με τον οποίο ε, ε εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Είχε ήδη, έχει ήδη διακοπεί η Ολομέλεια σήμερα το πρωί. Δεν μπορώ να ικανοποιήσω το έτοιμά σας. Το σημειώνω και θα το διαβιβάσω καταλήλως. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπέι από τους λεπτό. Ο εμφύλιο Πόλεμο μένεται από το 1972 στο Μπουρουντί με ελάχιστε περιόδου ηρεμία. Η πλειοψηφία Χούτου και η μειονότητα Τούτσι διαπράττουν σφαγέ. Οι εθνοτικές μειονότητες συχνά είναι σε μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι υποδιαιρέσεις, οι διάφορες ε, δείχνουν ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια και δεν ε, υπάρχει και λύση. Χάρη στις ε, προσπάθειες του πρώην Προέδρου Γιώγια, που ήταν πρώην Τούτσι και προσπάθησε με τη συμφωνία της Ισαρούσα να έρθει σε συνεννόηση με τους Χούτου. Δυστυχώς επανήλθαν και να ζωπηρώθηκαν οι παλιές ε, εντάσεις και αντιθέσεις. Φαίνεται ότι ο τωρινός πρόεδρος θέλει να ε, παραμείνει στην εξουσία ενώ απαγορεύεται από το Σύνταγμα να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Υπάρχει κίνδυνος να χυθεί πολύ ε, αίμα και καταχράται η Ευρωπαϊκή Ένωση του δικαιώματος παρέμβασής της στα πράγματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά για την επίλυση μιας τόσο περίπλοκης σύγκρουσης που γίνεται τόσο μακριά από τον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει και άλλο διαδικαστικό θέμα. Θέλετε και πάλι να ζητήσετε διακοπή της Ολομέλειας. Βάσει του άρθρου που αναφέρατε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αν τώρα θέλετε να πείτε κάτι άλλο, ευχαρίστως. Μιλάμε για τον ίδιο κανόνα, για τον ίδιο άρθρο. Εάν 40 μέλη της Ολομέλειας σηκωθούν και ζητήσουν αναστολή διακοπή της συνεδρίασης, αυτό πρέπει να γίνει πριν τη συζήτηση, αλλά εν δεν υπάρχουν 40 τώρα μέλη. Αλλά εν έχετε το λόγο. Ο κανονισμός λέει ότι μπορεί να γίνει διακοπή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κυρία Πρόεδρε, αν το αποφασίσει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του Πρόεδρου ή κατόπιν ετήματος μιας πολιτικής ομάδας ή 40 μελών τη. Τέτοιου είδου πρόταση θα ε, ψηφιστεί ε, αμέσως. Αυτό έγινε ε, στις 12 το μεσημέρι και όχι τώρα πρόσφατα. Σας παρακαλώ πολύ να προβούμε στην, στη χρήση αυτής τη διαδικασίας. Köszönöm felvetését. Ευχαριστώ πολύ το αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω ότι αναφερόμαστε στον ίδιο κανόνα. Υπάρχουν 40 μέλη που στηρίζουν αυτή την εκδοχή. Παρακαλώ να ε, σηκωθείτε. The political group, not all 40. Yes, really. all not and, Madam President. political group, all, not and. Υπάρχει ή διαζεκτικό, κυρία Πρόεδρε, ή 40 μέλη ή πολιτική ομάδα. Νομίζω ότι βλέπετε το ίδιο όπως και εγώ, ότι δεν υπάρχουν 40 μέλη, ο πρόεδρος δεν το ζητεί. Παρακαλώ να ηρεμήσετε και να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ε, ζητώ από το αξιότιμο μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μου επιτρέψει να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Ελπίζω να μην με διακόψετε. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Αν υπάρχει τέτοιο αίτημα εκ μέρους πολιτική ομάδα να μα το πείτε. Ποιο υποβάλλει το αίτημα και εκ μέρου ποια πολιτική ομάδα. Έχετε το λόγο. Το είπα στην αρχική μου ε, παρέμβαση. Εκ μέρους του EFTD ζητώ να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημά μας. Ευχαριστώ. Επομένως, πιστεύετε ότι αν θορυβείτε και φωνασκείτε, θα εγκρίνουμε το αίτημά σας, χωρίς να μιλάει κάποιος υπέρ και κανείς κατά. Βεβαίως ε, είμαστε βιαστικοί, αλλά παρακαλώ να έχετε υπομονή. Ποιος θέλει να σχολιάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόκειται ε, για έλλειψη σεβασμού προς, την, ε, ε, προς το Κοινοβούλιο. Αν δεν ενδιαφέρει του αδέλφους η κατάσταση του Μπουρούντι, καλύτερα να εγκαταλείψουν το ημικύκλιο εδώ. Μιλούμε για μια πολύ σοβαρή κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν την ημερησία διάταξη. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το Μπουρούντι και το πόσο ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι εκεί. Αν δεν του ενδιαφέρει να σηκωθούν να φύγουν. Επομένω, η Πρόεδρος, το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι κάποιος κατά του αιτήματο διακοπής της συνεδρίασης. Είναι κάποιος υπέρ, θέλει κάποιος να μιλήσει υπέρ του αιτήματο διακοπής της συνεδρίασης. Έχετε χρόνο. Έχουμε χρόνο για μια δημοκρατική συζήτηση. Θέλετε να συνεχίσετε να φωνάζετε ή θέλετε μια δημοκρατική συζήτηση. Δίνω το λόγο και στους υπολείπους που τον έχουν ζητήσει. Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα γίνει ψηφοφορία όταν κηρύξω την έναρξη τη ψηφοφορία. Τότε θα ψηφίσουμε. Θέλει κάποιο λοιπόν πρώτα να επιχειρηματολογήσει κατά. Θέλει υπέρ ή κατά θέλετε να επιχειρηματολογήσετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ να έχετε υπομονή. Πολύ περισσότερη υπομονή από αυτήν που έχετε επιδείξει. Διότι η αξιότιμη κυρία έχει δίκιο. Δεν δείχνετε σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ζητώ να ε, σεβαστείτε τη διαδικασία. Σας ζητώ να σταματήσετε να φωνάζετε, να ε, είστε ευγενείς και να συμπεριφέρεστε με τρόπο αξιοπρεπή σύμφωνο με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Σας μιλάτε τόσο δυνατά που σας ακούω και χωρίς να έχετε ανάψει το μικροφωνό σας. Έχετε το λόγο. Okay. Are you running θα μου δώσετε το λόγο. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να αξιοποιήσετε κάθε δυνατή ευκαιρία να στρέψετε τα φώτα της προσοχής πάνω σας. Θέλετε να δείξετε ότι ο Πρόεδρος δεν κάνει καλά τη δουλειά σας. Περίμενα πολύ περισσότερα από αυτή την ομάδα. Ωστόσο αυτό που κάνετε εσείς σήμερα είναι αναξιοπρεπές. Σαν μικρά παιδιά ε, όταν γίνεται συζήτηση, έχουμε επίτροπο εδώ, έχουμε σοβαρή συζήτηση για σοβαρό θέμα και κάνετε σαν μικρά παιδιά. Ε, δεν δείχνετε σεβισμό στην κατάσταση. Συγγνώμη, δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν δείχνετε σεβασμό ω προ την κατάσταση στο Μπουρούντι, μια κατάσταση η οποία είναι πολύ σοβαρή. Ε, ο κόσμο πεθαίνει. Είναι δραματική η κατάσταση στη χώρα αυτή. Δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα. Σοβαρά μιλάτε. δεν ε, επιτρέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να βγουν συμπεράσματα, να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε. Δεν τρέπεστε. Ερωτώ, δεν τρέπεστε. Παραδεχτείτε Παραδεχθείτε το ότι είναι αναξιοπρεπές αυτό από την περιλευρά σας. είναι όνειδος. Σκεφτείτε λίγο, αποχωρήστε από, από την αίθουσα και σκεφτείτε για την αντιδημοκρατική σας ε, συμπεριφορά. Και αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορώ να σας στείλω. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε το αξιότιμο μέλος για τη συνεισφορή του στη συνεισφορά του στη συζήτηση. Πρόεδρε, συγγνώμη, άκουσα τον κύριο να μου λέει να ε, το βουλώσω. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να καταγραφεί. Olyan Πρόεδρος, εγώ δεν το άκουσα αυτό το βουλοσέτο, αλλά ε, αν εσείς το ακούσατε βεβαίως θα καταγραφεί. Και ε, θα γίνει η ψηφοφορία και θα αποφασίσουμε. Έχετε το λόγο καταρχήν εσείς. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο και αυτό το επιλέξαμε εμείς. Και σήμερα το πρωί αναβλήθηκε μια συζήτηση που ήταν ε, και είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους τους Ευρωπαίους. γνωρίζουμε τους κανόνες, οι οποίους εσείς έχετε καθορίσει. Και ο κανόνας λέει να επιλύσει ένας υπέρ, ένας κατά. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Άρα δηλαδή ζητώ τώρα από την Πρόεδρο να δρομολογήσει την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ψηφίσουμε, όχι τώρα, θα διακόψουμε για μισή ώρα και μετά θα ψηφίσουμε.